και θα συμπεριληφθεί στα κείμενα που θα έχουν εγκριθεί αύριο. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου που ε, αναφέρθηκε χθε ότι δεν θα προβάλλει αντίρρηση ε, στην απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί τα παρατήματα 1, 2, 4 του 179 του 2012 ως προς το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων η πράσινη και η ενωτική αριστερά προέβαλαν αντίρρηση. Σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού θα εγγραφεί για ψηφοφορία την Πέμπτη αυτό το θέμα. Αύριο στις 10 η ώρα λίγη η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, ενώ ε, στις 4 το απόγευμα για την κατάθεση προτάσεων για ε, ονομαστική ψηφοφορία κατά τμήματα και χωριστή. Ευχαριστώ για την ιδιαίτερη προσοχή που δώσατε σε αυτό το θέμα. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση πρόοδου του 2013 για την Αλβανία δηλώσει του